Ασία, στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Θα συνεδριάσουμε αύριο 8 Οκτωβρίου από τις 8.30 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 19 μέχρι τις 7 το βράδυ λύεται η συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.